κοινή συζήτηση συμφωνίες αλληλευτικής σύμπραξης σύσταση του κυρίου Βαλέσα βιώσιμη μεταξύ, δηλαδή συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Λιβερίας και μετά σύσταση του κ. Μάτο Συμφωνία Αλευτικής Σύμπραξης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαυριτανίας, Αλευτικές Δυνατότητες και Χρηματική Αντιπαροχή. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κ. Βαλέσα. Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη συμφωνία ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Λιβερίας μαζί με ένα πρωτόκολλο το οποίο ετέθησε ισχύ το Δεκέμβριο του 2015. Θα εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα από το, αυτή τη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε καλή σχέση με την Λιβερία. Αυτό και προς όφελος της Λιβερίας και προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη. Ήδη συνεργαζόμαστε μέσω πολυμερών συμφωνιών ε, όπως το, η Σύμβαση των Ηνωμένων για το Δίκαιο της Θάλασσας και επιπλέον η Λιβερία συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση παράνομης αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλίας. Η νέα συμφωνία θα μας δώσει ένα πλαίσιο για να λάβουμε υπόψη τις ε, προτεραιότητες της μεταρρυθμισμένης ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής και τις εξωτερικές της δράσεις προκειμένου να δημιουργήσουμε μια στρατηγική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβερίας. Ο βασικός ε, στόχος του πρωτοκόλου είναι να δοθούν ε, αλληλευτικές δυνατότητες σε ευρωπαϊκά αλληλευτικά σκάφη στα ύδατα της Λιβερίας. Ε, το πρωτόκολλο δίνει δυνατότητα ε, σε 34 σκάφη από την Ισπανία και τη Γαλλία να αλλιεύουν 6.500 τόνους το χρόνο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώνει 650.000 ευρώ το χρόνο 50% ε, για την πρόσβαση και 50% για την στήριξη της αλευτικής πολιτικής Λιβερίας. Στόχος επίσης είναι να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβερίας, να προωθηθεί ε, βιώσιμη, πολιτική βιώσιμη αλίας και ε, οι αλευτικοί πόροι της Λιβερίας να τη χάνουν λογικής εκμετάλλευσης προς όφελος και των δύο πλευρών. Ενθαρρύνω λοιπόν το Κοινοβούλιο να ψηφίσει υπέρ τη συμφωνίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε και κύριοι, μιλούσαμε εδώ για την εξωτερική διάσταση της ε, ευρωπαϊκής ε, αλληλευτικής πολιτικής και στηρίξαμε την αλλαγή στρατηγικής που θα έπρεπε να εξασφαλίσει, να δώσει περισσότερες εγγύσεις στο στόλο μας, μεγαλύτερη διαφάνεια και μια βελτίωση ε, των συνθήκων τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για και τρίτων χωρών. Το αλληλευτικό πρωτόκολλο με την Μαυριτανία ακριβώς αποδεικνύει ότι κάνουμε βήματα πρόοδου προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, η συμφωνία αυτή είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη και για τον Ευρωπαϊκό Στόλο και για τον πληθυσμό της Μαυριτανίας ε, που θα λάβει όχι μόνο χρηματοοικονομική ενίσχυση ε, για την πρόσβαση στα ύδατά της αλλά και ενίσχυση για την ανάπτυξη του αλευτικού τομέα της. Αυτή η καινούργια σύμβαση με την Μαυριτανία επιλύει ορισμένα κενά του, ρυθμίζει ορισμένα κενά του προηγούμενου πρωτοκόλλου. Για παράδειγμα, οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί τότε είχαν μειώσει τη δυνατότητα ε, πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατότητων που μας έδιναν. Ε, δεδομένου ότι μας ε, ε απέκλειαν από την αλίευση κεφαλόποδων. Ε, οι αλευτικές ε, ζώνες επίσης βελτιώθηκαν έτσι ώστε να βελτιωθεί η συνύπαρξη με τα μαυριτανικά σκάφη. Βελτιώθηκε επίσης η, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η υποχρέωση πρόσληψης μαυριτανών ναυτικών. Ε, αυτή τη στιγμή ε, εξαιρούνται οι χειριστές ε, μηχανισμών και αυτό βελτιώνει την κατάσταση. Ε, επίσης γίνεται μια ρύθμιση για τα άκρος μεταναστευτικά είδη και οι κανόνες που εφαρμόζονται για μας είναι πλέον ίδιοι με αυτούς που εφαρμόζονται για άλλες τρίτες χώρες ιδιαίτερα για τον τόνο. Σε ό,τι δεν αφορά τις, ε, περιόδους αλίευσης, ε, την περίοδο αλίευσης είναι τέσσερα έτη η διάρκεια της συμφωνίας. Μέχρι τώρα οι συμφωνίες ήταν μικρότερες διάρκειας και το πρόβλημα που προέρχεται ήταν ότι ε, ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύω, τη θέση ισχύ της συμφωνίας, αρχίζαμε να διαπραγματευόμαστε την επόμενη συμφωνία. Πολλές βελτιώσεις λοιπόν και για το στόλο μας και για τη Μαυριτανία. Έτσι θα βελτιωθούν οι σχέσεις μας και θα λυθούν κάποια προβλήματα που υπήρχαν στην προηγούμενη συμφωνία, στο προηγούμενο πρωτόκολλο και στη σχέση επίσης με το στόλο τρίτων χωρών που αλλιεύαν στα ίδια ιδέα. Από οικονομικής πλευράς οι συνθήκες, οι όροι είναι πολύ καλύτεροι σε ό,τι αφορά το, τη σχέση κόστους-οφέλους. Σε αυτό ιδιαίτερα συνεισφέρουν τα τεχνικά μέτρα. Το πρωτόκολλο αυτό ήδη εφαρμόζεται από τον Νοέμβριο του 2005 προσωρινά και πιστεύω ότι ήδη έχουμε ένα θετικό απολογισμό. Αν και στο τέλος του Μάη θα λάβει χώρα η συνεδρία της Μικτής Επιτροπής για να αναλύσει ακριβώς τις εξελίξεις και να προτείνει ενδεχομένω και βελτιώσεις. Μία από αυτές θα έπρεπε να είναι η δυνατότητα να, να ξανααλλιεύσουμε κεφαλόποδα σε μαυριτανικά ύδατα. Αυτή τη στιγμή πληρούνται οι προποθέσει για να ξαναρχίσει αυτή η δραστηριότητα. Ξέρουμε όμω ότι η Μαυριτανία διαφωνεί αυτή τη στιγμή και αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι πολύ δύσκολη η συμπερίληψη των κεφαλοπόδων. Όμως θα θέλαμε να γίνει μια προσπάθεια ε, στην μεικτή επιτροπή που θα λάβει η χώρα μέχρι το τέλο Μαΐου. Άλλη δυνατότητα ε, να είναι δυνατόν τα αλλιεύματα ε, να ξεφορτώνονται στη, σε ευρωπαϊκά λιμάνια στην Γκραν Κανάρια πιο συγκεκριμένα. Ε, η, αυτή τη στιγμή επιτρέπεται η εκφόρτωση να γίνεται μόνο σε μαυριτανικές εγκαταστάσεις. Πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν ε, να αλλάξει το σύστημα, να δοθεί μια εξαίρεση μέχρι ότου τουλάχιστον βελτιωθούν οι μαυριτανικές υποδομές στα λιμάνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον λόγο και ο Επίτροπος Βέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω στην κοινή συζήτηση για τη Συμφωνία Ελευθερικής Σύμπραξης και τα συνδεδεμένα πρωτόκολλα με τη Λιβερία και τη Μαυρετανία. Με αυτή την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές, τους κυρίους ε, Βαλέσα και Μάτο για τις εκθέσεις. Η Επιτροπή Σαλίας συστήνει το Κοινοβούλιο να συμφωνήσει και με τις δύο συμφωνίες. Να πω δύο λόγια τώρα για κάθε μια από αυτές τις συμφωνίες. Πρώτα για τη Λιβερία. Η ε, νέα συμφωνία σύμπραξη βιώσιμης αλίας με την Λιβερία ε, δεν είναι από τις μεγαλύτερες συμφωνίες μας εις ό,τι αφορά τις αλλιευτικές δυνατότητες και την οικονομική συμμετοχή. Είναι όμως πολύ σημαντική συμφωνία διότι διευρύνει το περιφερειακό σύστημα ε, συμφωνιών για αλλιεύση αλλιατών ε, στη Δυτική Αφρική για τέσσερα χρόνια και μέχρι και θα μπορούν ε, ε, στην ε, ζώνη αλληλείας να αλλιεύουν τα σκάφη μας 28 θυναλιευτικά γρηγρή 6 παραγαδιάρικα επιφανείας. Θα επεκταθεί και η γεωγραφική κάλυψη των αλλιευτικών δραστηριοτήτων χωρίς να αυξηθούν οι ικανότητες. Η συμφωνία αυτή με τη Λιβερία επίσης σέβεται απόλυτα την αρχή της βιωσιμότητας των αλληλευτικών δραστηριοτήτων και στηρίζεται στα πλέον πρόσφατα και καλύτερα βέλτιστα επιστημονικά δεδομένα την αρχή της διαφάνειας και μη διακρίσεων άλλων στόλων. Ε, υπάρχει και ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συμφωνία επίσης αποστέλει ισχυρό μήνυμα ότι η Λιβερία είναι ανοιχτή για επιχειρηματικές δραστηριότητες παρά τις δυσκολίες στη χώρα με τα ε, ε, το πρόβλημα με τον έμπολα πέρσι. Ε, είναι πραγματική σύμπραξη, δεν ανοίγει μόνο αλλιευτικές δυνατότητες για τον ενουσιακό στόλο και ευκαιρίες για τη Λιβερία, δημιουργεί και ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη του, ελιευτη, του τομέα της αλίας στη Λιβερία και καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Ε, θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι για να ενισχυθεί η παρακολούθηση, ε, εποπτεία και έλεγχος. Έτσι θα μπορέσει να ε, ελέγχει τις ελιευτικές δραστηριότητες όλων των στόλων στα ύδατα της χώρας αλλά και τα δικά της για τα σκάφη συγγνώμη. Πρόσφατες συζητήσεις με τις λιβερικές αρχές άνοιξαν το δρόμο για συμπληρωματική δράση στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης και συνεργασίας με τη Λιβερία ε, για να υπάρχει και τομεακή κάλυψη. Τώρα η διαδικασία αυτή είναι στα Σπάργανα, αλλά οι λιβερικές αρχές ζήτησαν πρόσθετη υποστήριξη για να βελτιώσουν το αλληλευτικό τους δυναμικό ε, να μπορέσουν επίσης να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις τοπικές αγορές και πιστεύουμε ότι αυτή η σύμπραξη θα είναι ε, μακροπρόθεσμη. Τώρα με την Μαυρετανία η συμφωνία αλλίασε με την Μαυρετανία είναι η μεγαλύτερη ε, συμφωνία σύμπραξης ε, με οικονομικούς όρους. Δίνει ελευτικές δυνατότητες μέχρι 98 ενωσιακά σκάφη από 11 κράτη-μέλη και έτσι είναι κέρια σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το στόλο της. Το νέο πρωτόκολλο είναι το αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων, είναι σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο πρωτόκολλο και μπορεί να θεωρηθεί υπόδειγμα για τις διαπραγματεύσεις στο μέλλον και άλλων συμπράξεων, συμφωνιών συμπράξεων με άλλες χώρες. Συνάδει απόλυτα με την εξωτερική διάσταση της μεταρρυθμισμένης ε, πολιτικής αλίας όπως ανέφεραν η Μάτο και Βαλέζα. Σέβεται την αρχή της ε, βιωσιμότητας και επιβεβαιώνει τις αρχές της διαφάνειας της του προτιμησιακής πρόσβασης για τον ενωσιακό στόλο και μη διακρίσεις μεταξύ ξένων στόλων. Το πρωτόκολλο θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει απόδοση από τις επενδύσεις και τα χρήματα των φορολογουμένων και θα υπάρχουν βελτιωμένες τεχνικές προϋποθέσεις. Θα υπάρχει καλύτερη ε, εφαρμογή της τομεακής υποστήριξης με περισσότερη αιρεσιμότητα. Τώρα το βασικό είναι να διασφαλίσουμε την ομαλή εφαρμογή του νέου πρωτοκόλου. Σας διαβεβαιώνω ότι η Κομισιόν θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγης την κατάσταση όλων των αποθεμάτων που καλύπτονται από το πρωτόκολλο για να, ε, ε, να, υπάρχει βιωσιμότητα στις δραστηριότητες. Θα ελέγξουμε αν η Μαυρετανία σέβεται τις αρχές της διαφάνειας και των μη διακρίσεων. Και αυτό είναι κρίσιμο για να ε, μπορεί να λειτουργεί ο νοσιακός στόλος κάτω από τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις ίσες με τον άλλον στόλων. Αυτό είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι πρόσφατα η Μαυριτανία ε, έπαιξε ε, ηγετικό ρόλο στην πρωτοβουλία άρσης των ε, ελλημάτων. με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσετε την, νομίζω ορισμένη από εσάς τη συνάντηση με τη χώρα αυτή που προβλέπεται τέλος Μαΐου και θα μπορέσουμε να την διεξαγάγουμε με βάση τα παλαιά και το νυν πρωτόκολλο. Θέλουμε όμως να θέσουμε στην Μαυρετανία τη δυνατότητα δημιουργίας ε, μιας νέας κατηγορίας βενθοπελαγικών ειδών γιατί έτσι θα μπορέσουν να ωφεληθούν οι τράτες που δεν μπορούν να ψαρεύουν χταπόδια και κεφαλόποδα λόγω της ε, κακής κατάστασης των αποθεμάτων. Επίσης θα συζητήσουμε τη δυνατότητα να χαλαρώσουν λίγο οι υποχρεώσεις ε, για τα σκάφη πελαγικών ειδών και τη μεταφόρτωση ε, των αποθεμάτων ε, αποκλειστικά ε, στο λιμάνι Νουαντιμπού. Ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να συζητήσουμε πάλι αυτές τις ελληνικέ συμφωνίες και προσβλέπω στην υποστήριξή σας το μέλλον για τις συμφωνίες αυτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Ε, τώρα θα ακούσουμε τους ε, διάφορους συζητητές των ε, επιμέρους κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο κύριος Σεμπαστιά για ένα λεπτό από την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή Ανάπτυξης ανισχύει δύο πράγματα σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες ε, Αλίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Πρώτον, η βιωσιμότητα βιωσιμότητα για να αποφύγουμε την υπερεκμετάλλευση που μπορεί να καταστρέψει και να αφανίσει ορισμένα από τα είδη. Δεύτερον, τα κράτη με τα οποία υπογράφουμε αυτές τις συμφωνίες ε, θα πρέπει να έχουν ωφέλη που να, τους βοηθήσουν, να τις να ξεφύγουν από την εξάρτησή τους, μέχρι τώρα εξάρτησή τους. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντική η ύπαρξη ρητρών ανάπτυξης που θα επιτρέπει σε αυτές τις χώρες να βελτιώσουν την ανάπτυξή τους και την κατάστασή τους, να γίνουν πιο αυτόνομες. Αυτές οι ρήτρε επίσης βοηθούν στον έλεγχο και της εξέλιξης της εφαρμογής και στη διαφάνεια αυτών των συμφωνιών. Γι' αυτό το λόγο χαιρόμαστε για την ύπαρξη αυτών των ρητρών στις συμφωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τώρα κύριος Μουρεσάνη ένα λεπτό από την Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η, συμφωνία αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λιβερία θα δώσει περισσότερε ευκαιρίε και προβλεψιμότητα στα σκάφη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον όλο βιομηχανικό κλάδο. Από την οπτική γωνία τη Επιτροπή του Προπολογισμού πρέπει να δηλώσω ότι ο δημοσιονομικό αντίκτυπο αυτή τη συμφωνία στα προγράμματα τη ε, Επιτροπή θα είναι 3,25 εκατομμύρια ευρώ στα πέντε χρόνια που θα, ε, που θα κρατήσει η συμφωνία για την πρόσβαση των ευρωπαϊκών σκαφών στα ύδατα της Λιβερίας είναι σημαντικό να εντοπίσουμε πριν και ο εισηγητής ότι οι, οι μισές από τις δυνατότητες θα δοθούν στην ε, Λιβερία για την στήριξη του δικού τη αλλιευτικού κλάδου. Ο μισό πληθυσμό της χώρας ζει στα εισπαράκτης περιοχές και ασχολείται με την αλλία. Είναι σημαντικό λοιπόν να επιτύχουμε το στόχο της ανάπτυξη, υπεύθυνη και βιώσιμη αλλιευτική δράσης, βεβαιωνόμενοι ότι ο κλάδος φτάνει στο πλήρε δυναμικό του. Το καθοριστικό στοιχείο για μένα θα είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων αυτών ώστε να βεβαιωθούμε ότι τα δικά μας τα χρήματα θα δαπανηθούν σωστά και ότι πραγματικά υπάρχει αλλαγή που συντελείται στην πράξη. Ευχαριστούμε κύριος Κοράο για ένα λεπτό από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από την σκοπιά της Επιτροπής Ανάπτυξης, η συμφωνία με τη Μαυριτανία και τη Λιβερία είναι ένα βήμα πρόοδου. Είναι χώρες οι οποίες προσπαθούν να ανασυσταθούν μετά από πόλεμο, λοιμούς, επιδημίες και παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων. Θετικές ενδείξεις έρχονται και από τις δύο χώρες με ε, την κατάργηση της δουλείας της, ε, των, βασανιστήριων, ε, των στη Μαυριτανία και την στήριξη της νόμιμης εργασίας στη Λιβερία. Βεβαίω θα πρέπει να κρυζωθεί η φτώχεια και η οικονομική ανισότητα, καθώς και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των γυναικών στις χώρες αυτές. Έχουν κοινού πόρους οι χώρες αυτές και τις ίδιες θάλασσες, τα ίδια νερά. Εφόσον λοιπόν έχουμε περιφερειακή αλληλευτική συμφωνία όπου να μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες της ευρύτερης περιοχής, θα έχουμε μια πραγματική επιτυχία σε αυτή την περίπτωση. Με τι συμφωνίε αυτέ στρεφόμαστε προ αναπτυσσόμενε χώρε που έχουν ανάγκη και από ανθρωπιστική βοήθεια και η δική μα νομοδότηση περιορίζεται στο να δώσει συνένεση ή όχι προ την σύναψη συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε αποφάσει που έχει ήδη λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε κυρία Γκαρδία Ζαμπάλ Ρουμπιάλ από την Επιτροπή Προπλογισμών για να μισή λεπτό. Nu este. Δεν είναι εδώ, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Μιλάν Μον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ τον Επίτροπο για την ε, πολιτική σύναψη αλευτικών συμφωνιών που είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τον στόλο μας αλλά και για την ανάπτυξη του ελευτικού τομέα σε τρίτες χώρες μέσω της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης. Σας ενθαρρύνω Επίτροπο, να συνεχίσετε στον ίδιο δρόμο. Οι συμφωνίε με τη Μαυριτανία και τη Λιβερία, παρόλο ότι είναι διαφορετικέ μεταξύ του, είναι και οι δύο σημαντικέ για τον ευρωπαϊκό στόλο, συμπεριλαμβανομένε και τι γαλλικέ από προέρχομαι. Ο τόνο είναι το βασικό είδο που περιλαμβάνει τη συμφωνία με τη Λιβερία. Ε, είναι μεταναστευτικό είδο, οπότε είναι σημαντικό να διαθέτουμε ένα ολόκληρο φάσμα συμφωνιών. Το πρωτόκολλο με την Μαυριτανία είναι από τα πιο σημαντικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βελτιωθεί σίγουρα σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή του, αλλά δυστυχώς μία ακόμα φορά εξαιρείται ο στόλος που αλλιεύει κεφαλόποδα. Η, στη, η συνεδρίαση της ε, ε, Μικτής Επιτροπής της Βρυξέλλες στις 30 και 31 Μαΐου θα ασχοληθεί με το θέμα ε, των μηχανότρατων ε, ε που καταψύχουν τα ψυγείων. Θα ήθελα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Μερλούκιο, θα ήθελα μέχρι τότε να έχουμε νούμερα για τα, για το συγκεκριμένο... για τα συγκεκριμένα είδη, ε, έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα στη Μικτή Επιτροπή. Ε, ο Ευρωπαϊκό ε, Στόλος αλλιεύει με βιώσιμο τρόπο στα ύδατά μα. Είναι ο πιο ελεγμένο στόλο στον κόσμο. Ελπίζω να μην δώσει η Μαυριτανία αλληλευτικέ δυνατότητε, σε άλλου τόλους τρίτων χωρών που ελέγχονται πολύ λιγότερο από του δικού μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Ρόντουστ για να μισή λεπτό. Οι, συμπράξη, οι συμφωνίες σύμπραξης ε, αυτές ε, είναι πολύ αποτελεσματικός ε, τρόπος εφαρμογής της μεταρρυθμισμένης κάλπο και εκτός Ευρώπης διεθνώς, ούτως ώστε να φροντίσουμε για την βιώσιμη ε, αλληλεία. Ε, όμως χρειάζονται σαφείς προϋποθέσεις βιωσιμότητας, ε, συνέπειας, διαφάνειας που θα πρέπει να εφαρμόζονται. Με τις δύο διμερείς ε, συμφωνίες Λιβερίας ε, Μαυρετανίας έγιναν δύο σημαντικά βήματα για τη μακροπρόθεσμα βιώσιμη αλλία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, με τη Λιβερία από το 2007 υπήρχε από το 2007 συμφωνία ε, ε, ε, υπάρχει τώρα νέα συμφωνία και αυτή θα βελτιώσει την αλληλεία επιτόπου συμβάλλοντας στην μάχη κατά της παράνομης αλίας. Το πρωτόκολλο της Μαυρετανίας είναι η πηξίδα θεωρώ για την αλληλευτική πολιτική εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. τονίζω ιδιαίτερα τις διατάξεις για τη διαφάνεια. Είναι καθοριστικές και για το μέλλον. Το πρωτόκολλο προδιαγράφει ε, την ε, ε, λειτουργία της συμφωνίας. Οι κανόνες διαφάνειας είναι απαραίτητοι για να διαπιστώσουμε πόσα ψάρια μένουν διαθέσιμα για τον ευρωπαϊκό στόλο χωρίς να αφαιρέσουμε από τους ντόπιου αλληλείς το προϊόν που χρειάζονται για την επιβίωσή τους. Αυτό είναι σημαντικό για όλες τις συνεργασίες. Τη συμφωνία την στηρίζω κύριο... Ευχαριστούμε ο κύριος Χόκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Οι συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβερίας και Μαυριτανίας ε, μας βρίσκουν σύμφωνους. Είμαι πεπισμένος ότι η σύμπραξη για τη βιώσιμη αλληλεία ε, είναι πολύ σημαντική για την συνοχή της αλληλείας δημιουργώντας ε, θετικές συνέργειες που αφορούν μη διακρίσεις, διαφάνεια κλπ. Όλα αυτά είναι θετικά και για το μέλλον. Μια παρατήρηση μόνο θα ήθελα να κάνω, μια έκκληση αν θέλετε. Όταν πρόκειται για την αλληλεία τόνου Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, ότι αλλιεύονται και πολλοί καρχαρίες και αν και οι καρχαρίες είναι επικίνδυνοι για τον άνθρωπο, παρόλα αυτά δεν πρέπει να επιτρέπουμε την ε, αλλιευσή τους. Ε, τους κόβονται ε, τα πτερίγια και μετά πετούν, πετώνται πάλι στη θάλασσα. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται απαγόρευση που πρέπει να προσθεθεί σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει σχετική διάταξη, θα ήθελα όμως να υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νικολάη Νουρίκα 1,5 λεπτό. Είναι μια ωφέλιμη συμφωνία αυτή με τη Λιβερία και για τα δύο μέρη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής, ε, τα εξή σημεία της. Καταρχήν, ο τρόπος με τον οποίο χορηγούνται άδειε αλίευσης με βάση αυτή τη συμφωνία. Η, ε, η απαγόρευση χορήγηση ιδιωτικών ειδημερών αδειών, κάτι που συμμορφώνεται με τους δικούς μας ε, κανόνες περί ε, καταπολέμηση παράνομη αλληλεία. Η Λιβερία έχει προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα ωφελήσει τον αλληλευτικό τομέα στη Λιβερία, θα δώσει προστιθέμενη αξία στον αλληλευτικό της κλάδο. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Λιβερίας ζει από την αλία. Καλωσορίζω τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, βοήθησε το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει, το ενέπλεξε συζητήσεις, ε, το ενημέρωσε, εξασφαλίστηκε η διαφάνεια. Είναι απόδειξη συν, καλής συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κυρία Νίριαντα για ένα μισό λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχουν στοιχεία και αρχές στις αλληλευτικές συμφωνίες εταιρικής σύμπραξης όπως το ότι η επισητιστική ασφάλεια της Μαυριτανίας είναι καθοριστικό θέμα, για παράδειγμα, λόγω της έλλειψης τροφίμων σε αυτήν την χώρα. Και αναγνωρίζεται ότι η ελευτική βιομηχανία θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα αυτή να επισητίζεται. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται να έχει δώσει τη δέουσα προσοχή στις ανάγκες της Λιβερίας και της Μαυριτανίας στις διαπραγματεύσεις για την πρόσθετη πρόσβαση των στόλων τους στα, διάφορα, στα ύδατα που καλύπτονται από τι συμφωνίες. Εδώ είναι σαφές ότι οι αλλοίς στην ε, Λιβερία δεν είχαν λόγο ε, στις διαπραγματεύσει της συμφωνίας αυτής. Και το ίδιο και με τις διαβουλεύσεις που έγιναν στη Μαυριτανία. Είναι δεδομένη η άποψη ότι εξαπατήθηκαν από τους Ευρωπαίους οι Λιβεριανοί και ότι το σύνολο των ποσών που προσφέρθηκαν δεν ε, ε αντιστοιχούν στις αλληλεκτικές δυνατότητες που δόθηκαν στον αριθμό των σκαφών που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ύδατα. Έτσι λοιπόν παράνομη και παράτυπη αλλοία θα εξακολουθήσουν γιατί χρειάζεται ένα πραγματικά νόμιμο σύστημα για να προστατεύσουμε τη μικρή κλίμακα σταχνική αλληλεία και να έχουμε βιώσιμη διαχείριση των πόρων. Η εξωευρωπαϊκή στόλη ε, επίσης δεν ε, ρυθμίζονται μέσω της συμφωνίας αυτής διότι τα παραγαδιάρικα τεράστιων διαστάσεων έχουν πρόσβαση και ε, το αλληλευτικά αποθέματα της Λιβερίας δεν προστατεύονται ήδη από τους επίσημους φορείς της χώρας κατά αυτόν τον τρόπο. Πράγμα που συμβαίνει και σε άλλες τρίτες χώρες. Engstrom, 1 30 λεπτό η κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η συμφωνία αυτή, πενταετής, με βρίσκει σύμφωνη γιατί φροντίζει για μεγαλύτερη διαφάνεια και στήριξη του τομέα κέρια σημασίας για να αναπτύξει δικό της δυναμικό η χώρα. Όμως η υποστήριξη ε, μπορεί να βοηθήσει τη Λιβερία να στηρίξει την παράκτη αλληλεία, να αναπτύξει επιστημονικές μεθόδους και να ενισχύσει την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Προκειμένου περί της διαφάνειας, η συμφωνία είναι η καλύτερη από τις δύο. Ε, δηλαδή ε, σε σχέση με εκείνη της Μαυρετανίας. Θα πρέπει να δημοσιεύεται ε, κάθε συμφωνία, δημόσιες και ιδιωτικές συμφωνίες θα πρέπει να δημοσιεύονται. Η Λιβερία ήταν υποδειγματική επί σειράν ετών, το έκανε αυτό. Ε, μπορέσαμε να δούμε το παράδειγμα αυτό και ελπίζω να είναι πλήρης και αξιόπιστης οι πληροφορίες. Η συμφωνία της με τη Μαυρετανία είναι καλή από πολλές απόψεις. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί έτσι να αναβαθμίσει τα πρότυπα ε, και σε σχέση με άλλους θόλους Κίνα, Ταϊβάν, Ρωσία. Η Μαυρετανία υποσχέθηκε να, να δημοσιεύσει όλες τις συμφωνίες για καλύτερη διαφάνεια ε, και καλύτερη διαχείριση των ελιευτικών πόρων. Ε, θα πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη επίσης ε, τα θέματα υποστήριξης του ντόπιου πληθυσμού. Κύριε Σκόμπερν, χαίρομαι που σας βλέπω εκεί στην, στην, του Πρόεδρου. Ε, και άλλος ένας ε, μήνας ε, που σπαταλάμε λεφτά για να έρθουμε εδώ πέρα στο Στρασβούργο να συνεδριάσουμε. Α, και άλλη μια αληθική συμφωνία, μάλιστα δύο θα έλεγα. Μια καινούρια με τη Λιβερία, μια καινου, ανανεωμένη με τη Μαυριτανία. Και άλλη μια προδοσία των καθημερινών ανθρώπων. Αυτές οι συμφωνίες ε, αποτελούν ε, ε, ευρωπαϊκή κυριαρχία πικιοκρατία σε τρίτες χώρες. Και τους κλέβουμε τα ψάρια για να μπορούν να ψαρεύουν οι ίδιοι. Πόσοι Αφρικάνοι δεν γίνονται πιο φτωχοί. Πόσα χρήματα Ευρωπαίων φορολογούμενων πραγματικά πηγαίνουν για να τους βοηθήσουν, να βοηθήσουν τους καθημερινούς ανθρώπους υπάρχει μια παροιμία που λέει δώσε στον άνθρωπο ένα, σε, σε κάποιον ένα ψάρι και θα φάει μια μέρα. Μάθε του να ψαρεύει και θα τρώει σε όλη τη ζωή. Δεν το κάνουμε όμως. Του παίρνουμε το ψωμί του, τα ψάρια του, του το κλέβουμε και ε, ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή δυστυχώς συνεχώς και του παίρνει και το μικρόφωνο. Ε, δεν είναι αργά να μετανοήσετε. Ο κύριος Λεμπρετών έχει το λόγο. Merci, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από το 1989 υπογράφει αληθικές συμφωνίες με τη μαυριτανια Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία συμφωνία υπογράφηκε στις 10 Ιουλίου 2015 και θα έχει τετρατή διάρκεια. Είναι καλή συμφωνία διότι επιτρέπει στα ευρωπαϊκά σκάφη να πάνε να αλλιεύσουν στα νερά της Μαυρετανίας με σεβασμό των ε, όρων ε, ε, γιατί επιτρέπουν λοιπόν την αλίευση στα ευρωπαϊκά έδατα. 47.000 τόνοι από τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με 30.000 τόνους της περασμένης συμφωνίας και με αύξηση του ποσού. Όμως η Μαυριτανία είναι μια χώρα φτωχή, πρώτη στην ε, κατάταξη ε, του ανθρώπινου βιωτικού επίπεδου. Έτσι τα 4.250.000 ε, ευρώ παραπάνω που θα δοθούν ε, δεν αρκούν σε σχέση με το προηγούμενο ποσό. Και επίσης ε, είναι μεγάλο το ποσοστό των αλλιέων και ερναυτικών μεταξύ της, του πληθυσμού της Μαυριτανίας. Είναι μια συμφωνία η οποία εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σεβόμενη σε ένα βαθμό και τις ανάγκες της Μαυρτανίας. Ελπίζω να είναι ένα ορόσημο στην εξέλιξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μαυριτανία Γερμανία, κάτι που έλειπε τα τελευταία χρόνια και το εύχομαι για δύο βασικού λόγου. Πρώτα απ' όλα διότι ω Γάλλο η Μαυριτανία είναι μια χώρα γαλλόφωνη που βρίσκεται στη σφαίρα επιρροή τη Γαλλία. Και ε, έχω πάει εγώ ίδιο εκεί, ε, αποσπασμένο επισήμω από το γαλλικό κράτο και ξέρω επίση ότι και για τη συλλογική μα ασφάλεια το κράτο αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένα υποδειγματικό ε, σύμμαχο για την καταπολέμηση τη ε, ακραία ε, Ισλαμιστική τρομοκρατία. Θέλουμε λοιπόν ένα τέτοιο αξιόπιστο σύμμαχο να τον έχουμε κοντά μα. Ευχαριστούμε ο κύριος Σεράο για ένα μισό Θέλω και εγώ να συγχαρώ τους ε, εισηγητές καταρχήν. Ε, ως ο εισηγητής εκ μέρους των Συνελτών και Δημοκρατών για τη συμφωνία με τη Λιβερία με ανησυχεί λίγο το θέμα της διαφάνειας. Για το κατά πόσον η Λιβερία σέβεται τις ε, αρχές Ευρωπαϊκής Ένωση μεταξύ αυτών της, ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων πώς, τι ποσοστό της βοήθειας ε, θα αφιερωθεί στην, στο σεβασμό των περιβαλλοντικών επίσης ε, ε, αρχών. Η Λιβερία μετά από δύο εφηλίους πολέμους και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς η οικονομία της Λιβερίας αρχίζει και ανακάμπτει σιγά σιγά. Ε, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να την υποστηρίξουμε, γιατί είναι η πρώτη συμφωνία της Λιβερίας. Για αυτή τη χώρα που βρίσκεται σε αναδιάρθρωση και ανοικοδόμηση είναι σημαντικό να δώσουμε κίνητρα και να εντείνουμε τις σχέσεις μας, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Και οι δύο συμφωνίες αλίας και με τη Λιβερία και με τη Μαυριτανία επιτρέπουν την αύξηση των ελευτικών δυνατοτήτων για τον ε, ευρωπαϊκό ελευτικό στόλο για την εκμετάλλευση, βιώσιμη εκμετάλλευση ελευτικών πόρων που δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές οι χώρες. Ε, επίσης ε, βελτιώνουν την ε, τροφιμική ασφάλεια στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο τις υπερψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στηρίζω την σύναψη αυτών των συμφωνιών. και για συναισθηματικού λόγους και για λόγους λογική. Ε, είμαι από οικογένεια ναυτικών και χαίρομαι για τη χαρά που δίνουν αυτές οι συμφωνίες τους ε, αλληλείς της περιοχής μου, της χώρας μου, της πόλης μου. Είναι ένας τομέας δύσκολος, ένα κλάδος πολύ δύσκολος και πράγματι θα πρέπει ε, να χαίρουν το σεβασμό μας όλοι αυτοί οι ναυτικοί και οι αλίες. 124 αλλιευτικά σκάφη από την Ευρώπη θα μπορέσουν να αλλιεύουν σε αυτά τα ύδατα των δύο χωρών. Όμως δεν θα είναι μια απλή αλλία, θα είναι βιώσιμη αλλία σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και χωρίς άναρχη και παράνομη αλλία. Θα ωφεληθούν και οι τοπικές κοινότητες και Τέτοιου είδου συμφωνίες νομίζω ότι ωφελούν όλα τα μέρη. Ανοίγουμε δρόμο με τη Λιβερία, ενώ με τη Μαυριτανία επαναλαμβάνουμε και βελτιώνουμε μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες. Θα πρέπει να λύσουμε το θέμα των κεφαλοπόδων όμως, πολύ σημαντικό για τα Κανάρια. Όμως ε, διατηρούμε τον έλεγχο των λευτικών διαδικασιών και την ε, ε, και την οικονομική στήριξη των χωρών αυτών. Ε, είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε αυτές τις συμφωνίες να αντισταθούν από άλλες λιγότερο βιώσιμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για τη δουλειά του και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον για τους εισηγητές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συμφωνίες εταιρικής σύμβεψης πρέπει να έχει τις ίδιες αρχές και πρότυπα που εφαρμόζονται και στα ευρωπαϊκά είδατα. Αυτό είναι δίκαιο. Όταν αλλιεύει κανεί τα νερά και τα είδατα τρίτων χωρών, θα πρέπει να υπάρχει και απαραίτητη υποστήριξη στην τοπική αλλία για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή ε, εμπλεκόμαστε θετικά με χώρε που έχουν ανάγκη από αυτού του τη στήριξη και καθημάς ε, κατανομή ευθυνών μεταξύ Ευρώπη και τρίτων χωρών πρέπει να γίνει ένα στόχο προτεραιότητα. Γι' αυτό εκτιμούμε τι εργασίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά στο να προβλέψει τέτοιου είδου συμφωνίε και κριτήρια. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να εξακριβώνουμε και να παληθεύουμε πριν τη σύναψη συμφωνία ότι οι αρχέ που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανταλλαγή αλληλευτικών δικαιωμάτων όντω θα ωφελήσει του τοπικού πληθυσμού το όντι, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στο γεγονός ότι οι μεγάλοι στόλοι μας με βιομηχανικές δυνατότητες ε, αποψηλώνουν από τους πόρους τους αυτά τα ύδατα και οι τοπικοί πληθυσμοί μπορεί να γίνονται πιο φτωχοί. Κλείνω. Λέγοντα ότι οι συμφωνίε αυτέ ελπίζουμε ιδίω για τη Λιβερία που είναι κράτο σε κατάσταση ανόρθωση να μπορέσει όντω να ωφελήσει. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αγγιγέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τους δύο εισηγητές ε, για τα αποτελέσματα αυτών των συμφωνιών. Πολύ σημαντικές ε, για τον Ευρωπαϊκό Στόλο και ιδιαίτερα για τον Ισπανικό Αλλιευτικό Στόλο. Χαίρομαι λοιπόν και στηρίζω τη σύναψη αυτών των συμφωνιών με τη Λιβερία και τη Μαυριτανία. Πιστεύω ότι ε, οι συμφωνίες βελτιώθηκαν, είναι βελτιωμένες σε σχέση με προηγούμενες συμφωνίες. Μπαίνουν ε, λοιπόν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και οι συμφωνίες αυτές είναι σημαντικές και για τον Ευρωπαϊκό Ελευτικό Στόλο ε, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Λυπάμαι που δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κεφαλόποδα μεταξύ των ειδών τα οποία θα μπορούν να λιεύουν οι στόλοι μας. Κρίμα, διότι τα κεφαλόποδα υπήρχαν στο προηγούμενο πρωτόκολλο και τώρα εξαιρέθηκαν. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να εισαχθούν στο μέλλον, μάλλον όχι, αλλά είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε. Στην επόμενη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής, 30 και 31 Μαΐου, θα αναλυθεί η ε, συμπερίληψη των, ε, παρα, των ε, μηχανότρατων ψυγείων. Είναι σημαντικό να, το, να τις προσθέσουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Μπλάνκο. Η σύναψη διεθνών συμφωνιών αλίας είναι πάντα καλή είδηση. Οπότε είναι καλή είδηση που καταλήξαμε σε αυτές τις συμφωνίες με την Λιβερία και τη Μαυριτανία. Είναι καλή είδηση για τον Ευρωπαϊκό Αλλιευτικό Στόλο. Μιλούμε για παραπάνω από 120 αλλιευτικά σκάφη της Ευρώπης, αλλά είναι και καλή είδηση για την ανάπτυξη των δύο αυτών χωρών με τις οποίες συνάπτουμε συμφωνίες. Θετικό βήμα λοιπόν. Δεν θα επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα και εγώ η συμφωνία με τη Μαυριτανία να έχει συμπεριλάβει και τον σκάφο κεφαλοπόδων και το στόλο κεφαλοπόδων, συγγνώμη, που είναι πολύ σημαντικός για τη Γαλλικία. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν να ενώσω τη φωνή μου με τους άλλους συναδέλφους και να ζητήσω αν είναι δυνατόν να διεκδικηθεί αυτό στο μέλλον και να σας ε, ενθαρρύνω κύριε Επιτροπέ να εργαστείτε προς την ίδια κατεύθυνση για καινούριε αλληλευτικές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στη διαδικασία ΚΑΤΣ ΚΑΤΣ-ΔΙΑΗ. Ο κύριος Μπόκοβιτ πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είμαι από θαλάσσιο κράτος που θα ωφεληθεί από την Ελία στα Αφρικανικά ύδατα, αλλά παρόλα αυτά συμφωνώ με τις δύο συμφωνίες για έναν απλό λόγο. Όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως και οι συγητές θεωρώ ότι φροντίζει για δύο πράγματα η συμφωνία. Αφενός ε, τον Ευρωπαϊκό Αλλιευτικό Στόλο και ε, παρέχει και αναπτυξιακή βοήθεια σε αυτές τις χώρες Αυτές είναι αφρικανικές χώρες που υπέφεραν πολλά δεινά λόγω διαφορετικών προβλημάτων όπως ασθένειες και άλλα ε, προβλήματα και πιστεύω ότι όταν συζητούμε κάθε μία από αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει να εξασφαλίζουμε υψηλή ανθρωπιστική βοήθεια που είναι το περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε για τις χώρες αυτές αφενός και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αφετέρου βάλει στη δημιουργία θέσεων εργασία σε πολλέ χώρε εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εύλογη εξωτερική αλλιευτική πολιτική τη Ένωση, οφείλει να διασφαλίζει τα συμφέροντα των ευρωπαίων αλλιέων ιδιαίτερα των μικρότερων να επιτάσσει την βιωσιμότητα την διατροφική ασφάλεια και την καταπολέμηση τη παράνομη αλλιείας εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώ οι συμφωνίε αλλιευτική σύμπραξη Ευρωπαϊκή Ένωση, λιβερία και μαυριτανία οφείλουν να περιλαμβάνουν σαφεί ρήτρε για την προστασία των αλλιευτικών αποθεμάτων την καταπολέμηση της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλληλεία αλλά κυρίως κύριε Βέλλα, τον σεβασμό θεμελιωδών εργατικών δικαιωμάτων στις δραστηριότητες των αλλιέων στις χώρες αυτές. ιδιαίτερα πρέπει να επισημάνουμε ότι η μαυριτανία είναι μια χώρα όπου υφίσταται κύριε Βέλλα, καθεστώς δουλείας για 150.000 ανθρώπους της φυλής χάρατιν ήτι το 4% του πληθυσμού. αυτό είναι απαράδεκτο και η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να καταδικάσει και να αποφύγει πλέον καμία, κάθε συμφωνία με τη μαυριτανία. Τι έχετε να πείτε για αυτό το θέμα κύριε Βέλα; Θα υπογράψετε αλλιευτική συμφωνία με τη Μαυριτανία όπου υπάρχει δουλεία. Περιμένω κύριε Επίτροπε μια απάντηση για το θέμα αυτό. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Βέλα. Καταρχήν συγχαρητήρια στους δύο συναδέλφους Μάτο και Βαλέσα που έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Οι συμφωνίες σύμπραξης με τις τρίτες χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τώρα αναβαθμίζονται ποιοτικά και μαζί με την Κομισιόν πιστεύω και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ε, παραγνωρίσουμε ότι τα, τα ψάρια είναι γενικό αγαθό ε, απαραίτητο για τον επισητισμό διεθνώς οι χώρες που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τους πόρους τους για διάφορους λόγους, γιατί είναι μικροί στόλοι, γιατί δεν έχουν τις σωστές τεχνολογίες. Με αυτές τις χώρες λοιπόν όπως Λιβερία, Μαυρετανία συνάπτουμε συμφωνίες που έχουν ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο. Δηλαδή όταν οι, ε, καταβάλλονται οικονομικές αντιπαροχές για την ανάπτυξη της αλληλείας σε μικρής και μεσαίας κλίμακας, για να μπορούν οι άνθρωποι ε, να, να παράγουν εισόδημα και διατροφή. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και νομίζω ότι αν θέλουμε βιώσιμη αλληλεία με βάση το βασικό κανονισμό μας, ε, αν, ε, θα, ε, θα πρέπει, ε, θα πρέπει να φροντίσουμε τις συμφωνίες αυτές και όχι να τους αφήνουμε σε άλλες χώρες που δεν τηρούν τις συμφωνίες όπως η Ρωσία εκείνη. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Πίτροπος, ο κύριος βέλε. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές για τα σχόλιά τους και τις συνεισφορές τους. Ω προ τη Συμφωνία εταιρική Σύμπραξη για τη Βιώσιμη αλήθεια είναι σημαντικά βήματα πρόοδου. Για του εξή λόγου. Πρώτα απ' όλα η συμφωνία με τη Μαυροτενία είναι μέχρι τώρα η μεγαλύτερη. Η συμφωνία με τη Λιβερία θα φέρει ε, εισοδήματα αληθικά και θα στηρίξει του αλήθειε σε μια χώρα που ακόμη προσπαθεί να επιβιώσει από το περσινό κρούσμα και το ξέσπασμα του Ιουέμπολα. Έτσι όλα τα μέρη, όλες οι πλευρές θα ωφεληθούν κατέρευθεν από την παρακολούθηση, τους ελέγχους και την ε, ε την ε, βιωσιμότητα και τις περισσότερες συμφωνίες που αυτό μπορεί να επιφέρει θα ε, ε, υπάρξει ε, αντάλλαγμα για το χρήμα που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Και εδώ οι συμφωνίε αυτέ στηρίζονται και από το σώμα σα, από ό,τι φαίνεται. Να κάνω λοιπόν κάποια συγκεκριμένα σχόλια. Υπήρξαν κάποιοι συνάδελφοι, Σεμπάστια, Μπριάνο, που ε, αμφισβήτησαν την βιωσιμότητα των συμφωνίων αυτών. Ναι, οι συμφωνίες εταιρική σύμπραξη, βιώσιμη αλίας που συνάπτονται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ε, των χωρών αυτών είναι ένα πραγματικά ιδιαίτερα ρυθμισμένο πλαίσιο για το πώ αλλιεύει ο Ευρωπαϊκό Στόλο στα ίδια των τρίτων χωρών. Είναι ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ελεκτικέ δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Στόλου γίνονται σεβαστέ και σέβονται το κατάσταση των αποθεμάτων, τι ανάγκε τη βιοπικιλότητα και τα οικοσυστήματα των χωρών αυτών και ότι δεν ανταγωνίζονται ούτε πλήττουν του ντόπιου αλλή. Είναι υπόδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε και κανένα άλλο στόλο ε, δεν έχει κάνει αντιστοιχό δίχω κάτι ανάλογο για την διαφάνεια και την καλή κυβέρνηση σε τρίτε χώρε και στα νερά των χωρών αυτών. Άλλοι, μιλάνμονα, Μόνα, Γκιλέρα, Μπλανκολόπε, Σποκ, ε, μίλησαν για τα κεφαλόποδα. Εδώ πρέπει να πω ότι τα πιο πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα δείχνουν ότι τα ανάλογα αποθέματα υπεραλλιεύονται. Επιπλέον η Μαυριτανία επιβεβαίωσε στην πράξη την πρόθεσή της να ε, διατηρήσει αυτό το αλλιεύμα για τον τοπικό της στόλο, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πλεόνασμα ούτε ηλιευτικέ δυνατότητε. Δεν μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε τέτοιε. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει άκοπα τι διαβουλεύσει με τη Μαυριτανία προκειμένου να εγκριθεί ένα σύστημα μέτρων βιώσιμη διαχείριση για να ανακτηθούν τα αποθέματα αυτά. Επίσης έγινε μια μνήα για τους καρχαρίες, νομίζω ο κύριος ε, Πόκτο ανέφερε αυτό, για τους καρχαρίες και εδώ πρέπει να πω ότι ο στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, αλλιεύει καρχαρίες, ούτε κάνει τέτοια πράγματα στους καρχαρίες, είτε εντός είτε εκτός ευρωπαϊκών υδάτων. Ένας αριθμός βουλευτών επίσης ανέφεραν τους ε, στόλους τεχνικής αλίας, μικρής κλίμακας. Αυτός ο τομέας στηρίζεται και στις δύο χώρες, ε, καθώς είναι σημαντικός ε, για την ανάπτυξη των χωρών αυτών, και της μικρής κλίμακας και της ερασιτεχνικής αλίας. Και για τη Λιβερία και για τη Μαυριτανία, οι συμφωνίες αυτές όχι μόνο θα εξυπηρετήσουν τον ευρωπαϊκό στόλο, αλλά και τις χώρες αυτές τις ίδιες. Θα μπορέσουν και αυτές ε, αν όλα πάνε καλά, να ε, λύσουν κάποια από τα κοινωνικά τους προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βαλέσσα για δύο λεπτά. Uh, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη συμβολή στη συζήτηση απόψε. Κάθε φωνή είναι σημαντική γιατί δίνει πρόσθετη συμβολή σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με αυτές τις μοναδικές και βιώσιμες συμφωνίες με τις χώρες αυτές. Επιθυμώ μόνο κάποια στιγμή σε κάποια συζήτηση για την Αλία να γίνει συζήτηση ε, κάποιο πιο λογικό χρονικό διάστημα και όχι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Μάτο, δύο λεπτά. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους παρενέβησαν. Αύριο θα ψηφίσουμε μια συμφωνία που, ε, της οποίας διαπραγμάτευση ήταν πολύ δύσκολη. Όμως το αποτέλεσμα πολύ θετικό. Η Μαυριτανία είναι μια χώρα με πολλές ανάγκες, αλλά όπως και πολλές άλλες χώρες Αφρικής είναι μια χώρα με πολλές δυνατότητες, πολύ δυναμικό και θα πρέπει να συσφίξουμε τη σχέση μας μαζί της. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εδώ και πολλά χρόνια στα Κανάρια με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσουμε διμερεί προγράμματα με τη Μαυριτανία πολύ ενδιαφέροντα όπως το Μακαπέλ πολύ πρόσφατα που δίνουν, ανοίγουν ορίζοντες και για τις δύο πλευρές. Ε, από ό,τι φαίνεται έχει κλείσει η δυνατότητα εκφορτώσει να γίνονται στα Κανάρια. Ε, ε, έτσι είναι σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πρέπει να υποχωρήσουμε, θα πρέπει να επιμείνουμε. Θα πρέπει να επιμείνουμε γιατί οι εκφορτώσει στα Κανάρια όχι μόνο είναι εύκολο να γίνουν, αλλά δεν βλάπτουν κιόλα την Μαυριτανία. Οπότε θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό μας το αίτημα. Ε, μην υποχωρείτε. Ε, το πλαίσιο είναι καλό και μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο για τις μελλοντικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση διαφάνειας με όλες τις διμερείς συμφωνίες. Τέλος, σας ζητώ την υποστήριξή σας προκειμένου να υιοθετηθεί αυτή η σύσταση και θα ήθελα ήδη να ευχαριστήσω την Κομισιόν και όλους εδώ στο Κοινοβούλιο που προσπάθησαν για πολύ καιρό να καταλήξουμε στην πιο ωφέλιμη, στην πιο θετική συμφωνία που μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται η κοινή αυτή η συζήτηση.